Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Γκαρντίνη με θέμα «Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των καταστροφών, ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας». Θα αρχίσουμε την συζήτηση με την εισηγήτρια. Κυρία Γκαρντίνη, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω